ασκούν μη βιώσιμη αλεία. Θα πρέπει και εμείς να εφαρμόζουμε τις ίδιες προδιαγραφέ και να είμαστε το ίδιο απαιτητικοί και με τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ε, έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι και το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η έκθεση της ε, Κορατσαμπίλτ, Άννα Μαρία Κορατσαμπίλτ, εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ε, η κατάσταση και τα επόμενα βήματα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κορατσαμπίλτ. Τέσσερα λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, στην Ευρώπη, χωρίς όμως να σπαταλήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Η οδηγία για τις υπηρεσίες ε, υπάρχει στα στόματα όλων μας από το 2006, όμως ε, κυρίες και κύριοι να μην ενδώσουμε στην κόποση που αφορά αυτή την οδηγία. Το θέμα που τίθεται είναι πώς θέσεις απασχόλησης χάνονται καθημερινά, γιατί δεν λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά. Ε, για την παροχή υπηρεσιών. Ε, Διερωτώ μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι περίπου το 70 80% ε, της οικονομίας, ε, πυλώνας της οικονομίας έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά όχι αρκετά γρήγορη και εξακολουθούν να υπάρχουν αδικαιολόγητοι φραγμοί που παρεμποδίζουν την ε, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί σε αρκετά κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε πρέπει να αντιρωτηθούμε κατά πόσο είναι σωστό ένας αρχιτέκτονας που θέλει να ε, εγκατασταθεί σε μια άλλη χώρα, κατά πόσο πρέπει να υφίσετε περιορισμού ή όχι. Να υπάρχουν <clears throat> ακριβότερες τιμέ για μη κατοίκου, Κύριε Πρόεδρε, ε, θα πρέπει να αποκτήσετε και άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο όταν έχετε ήδη το δικό σας ε, στην πατρίδα σας. Αυτό είναι απαράδεκτο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω την πολύ καλή δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως την προσωπική αφοσίωση του κυρίου Μπαρνιέ, σας καλωσορίζω κιόλας, ε, για την πολιτική μη ανοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει παραβιάσει και το ε, Οκτώβρη θα ενημερώσει το Συμβούλιο για περιορισμούς ε, με στόχο να μεγιστοποιηθεί ε, το οικονομικό όφελος. Ξεκολουθούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχουν κανόνες, όμως αυτοί δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε τη διαδικασία επιπαραλήψη που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ ε, κάποια κύρωση, κάποια τιμωρία. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Ιρλανδική και τώρα και με τη Λιθουανική Προεδρία και τα θέματα αυτά θέλουμε να τα βάλουμε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Θέλω επίσης να απευθυνθώ στα Εθνικά Κοινοβούλια και σε όλους τους εμπλεκόμενους να τους καλέσω να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν πλήρω την οδηγία παροχή υπηρεσιών. Καλή την πίστη βέβαια. Αυτό όμω δεν αποτελεί ε, δικαιολογία. Εξακολουθούν να είναι υπόλογοι στου ε, Ευρωπαίου πολίτε. Πρέπει να άρουμε του φραγμού, γιατί αυτό είναι ένα αποτελεσματικό τρόπο για να προκαλέσουμε ανάπτυξη. Και πιο συγκεκριμένα κύριε Πρόεδρε πρέπει να δούμε λιγάκι τι γκρίζε ζώνε, την κατάκνηση και την ανασφάλεια που προκαλούν σύγχυση σε όσους προσφέρουν υπηρεσίε. Ε, εδώ λοιπόν ε, αναφέρομαι στις εθνικές αρχές ε, και απευθύνομαι σε αυτούς ε, να τους ε, πω ότι πρέπει να κάνουν ε, τις παρέτητες αξιολογήσει. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για το πώς θα εφαρμόζουν τα τεστ αναλογικότητας. Επίσης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στην αξιολόγηση ομοτήμων θα πρέπει να μεριμνούμε έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών. Μία προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν παρεμβάσεις από άλλα κράτη-μέλη. Η πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο που θα είναι γνωστός σε όλους. Και το πιο σημαντικό από όλα κύριε Πρόεδρε και τελειώνω με αυτό, νομίζω ότι η εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών πρέπει να συμπεριληφθεί στην, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και να παραμείνει εκεί για όσο καιρό χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Μπαχνιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση για πολλούς λόγους. Είναι πολύ καλή η έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλ, την έκθεση την οποία έχει διαμορφώσει με, την συνήθη, με τον συνήθι ενθουσιασμό της και η κυρία Γκέπχερτ και η κυρία Σλίξ στη συνέχεια ε, δούλεψαν πάνω σε αυτό τον τομέα των υπηρεσιών και αυτή η έκθεση τώρα συνεχίζει. Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία ε, Γοράτσα οι υπηρεσίε καλύπτουν ένα πολύ σημαντικό τομέα που έχει ένα τεράστιο δυναμικό ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση, μια στιγμή που τι χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. 45% των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτονται από την οδηγία αυτή και θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά η οδηγία. Αυτή η οδηγία δεν είναι το παν, πρέπει επίσης να, ε, να κινητοποιηθούμε ε, σε τομείς που βρίσκονται οριακά σε αυτήν την οδηγία ε, και που είναι σε αναδιάθρωση όπως είναι το λιανεμπόριο η κυρία Κοράτσα Μπίλτ το ανέφερε και αυτό και το online, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, θα αναφερθώ σε αυτή την έκθεση με βάση την ανακοίνωση που είχα κάνει τον Ιούνιο του 2012 για να υπενθυμίσω ότι είναι υψηλό το επίπεδο των απαιτήσεων για την υλοποίηση της οδηγίας αυτής. Καταρχήν, μηδενική ανοχή το κείμενο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί πλήρως και έχουμε θέσει στόχο την μηδενική ανοχή, πολύ αυστηρό κατόφλι για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη και υπό το πνεύμα αυτό έχουν ξεκινήσει προδικαστικές διαδικασίες ε, με κάποια κράτη-μέλη. Πέντε κράτη-μέλη mm. ήδη ε, συμμορφώθηκαν και η Επιτροπή συνεχίζει την επαφή με τα υπόλοιπα κρατημέλη για να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία εμένουν. Δεύτερον, ο τομέας των αποκαλούμενων επαγγελματικών υπηρεσιών. Το 2012 ξεκίνησε μια διαδικασία αξιολόγησης από τους ομοτήμους για να εμφανιστούν τα συστήματα τα οποία είναι λιγότερο περιοριστικά για την ε, ελεύθερη ε, παροχή υπηρεσιών. Και επί τη βάση αυτής της δουλειάς, σύντομα θα δημοσιεύσουμε ένα έγγραφο που αναφέρεται στα θέματα, σε νομικά θέματα και σε θέματα κεφαλαίου. Και θα καλέσουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μία επανεξέταση των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε χώρα. Τρίτον, η ενιαία ε, θέση παροχής πληροφοριών ε, με τόσες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται πραγματικά σπαζοκεφαλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσει το που πρέπει να απευθυνθούν ε, για να ε, ενημερωθούν. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ενιαία θηρίδα ε, που θα πρέπει να λειτουργεί και αποτελεσματικά. Προτείνω λοιπόν ένα χάρτη για τις ενιαίες θηρίδες που ε, θέτουν ε, νέα στάνταρ ποιότητα για μια δεύτερη γενιά κέντρων εξυπηρέτησης θηρίδων τέτοιων που μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το διαδίκτυο και θα υπερασπιστεί η Επιτροπή αυτή, αυτό το νέο θεσμό και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να θέσουν στην διάθεση των πολιτών τέτοιες θηρίδες για να εξυπηρετούν του πολίτε για την οδηγία για τι Υπηρεσίε. Τέταρτο σημείο, το άρθρο 20. Προστασία των καταναλωτών, όπω αναφέραμε και σε άλλη συζήτηση στην Ολομέλεια το πρωί, αποτελεί προτεραιότητα. Η προστασία των καταναλωτών καλύπτει ε, την επιθυμία των πολιτών να μπορούν να αγοράσουν εμπορεύματα ή αγαθά υπηρεσίες οπουδήποτε και αν είναι ο τόπος κατοικίας τους. Και ε, μία ανακοίνωση της Επιτροπής ασχολείται με την μη διάκριση, μη διακριτική μεταχείριση για την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων ε, online και ε, πολλές φορές συμμετέσχω και εγώ στη διαμόρφωση σχετικών μέσων και έτσι θα βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές με τα μέτρα τα οποία διαμορφώνουμε και ε, μέχρι το τέλη του έτους θα δημοσιεύσουμε και ένα έγγραφο προς ε, τους καταναλωτές και προς τις επιχειρήσεις όπου θα καταγράφονται τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν αγοράζουν κάτι από ένα άλλο κράτος μέλος. Λοιπόν, αυτή η δράση μα προχωρεί πέρα από την οδηγία για τι Υπηρεσίε, παρότι είναι προτεραιότητα για μα να εφαρμόσουμε όλα τα μέσα που θα δώσουν στην οδηγία αυτή το πλήρες δυναμικό της. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα σημείο που μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και όχι μόνο σε μένα. Ε, το θέμα αυτό είναι η κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των υπηρεσιών. Γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα των συζητήσεών σα. και συμφωνώ με τη δική σα άποψη ότι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών θα πρέπει να τίθεται στην ε, διάθεση όλων των επιχειρήσεων, των καταναλωτών αλλά και των μισθωτών ε, και άλλων εργαζομένων η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων ούτε να οδηγεί σε καταχρήσεις είτε σε αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών. Και η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ξεκάθαρη για το θέμα αυτό. Εξάλλου εσείς ε, έχετε πιστήσει την προσοχή στο θέμα αυτό όταν υιοθετήθηκε η οδηγία δεν θα πρέπει να θίγεται ε, το εργατικό δίκαιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης δεν θα πρέπει να θίγεται το δικαίωμα διαπραγματεύση, το δικαίωμα για συλλογικέ συμβάσει και το δικαίωμα σε συλλογικέ δράσεις. Δεν επηρεάζεται η νομοθεσία των κρατών μελών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης τούτου ε, λεχθέντος ε, θα πρέπει να εντείνουμε την ε, προσπάθειά μας για να αποφεύγονται οι καταχρήσεις σε θέματα απόσπασης εργαζομένων και σε θέματα απάτης στο φορολογικό τομέα. και εξετάζεται η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων ε, από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά ε, τους παρέχοντες υπηρεσίες ε, προσωρινή βάση, με την απόφαση λιμόζα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μιλά για το κράτος μέλος υποδοχής. Είναι σαφές ότι στην προσέγγιση του Δικαστηρίου αλλά και της Επιτροπής τα μέτρα τα οποία προτείνονται θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να ανταποκρίνονται στους στόχους, δηλαδή που είναι, ο στόχος είναι η καταπολέμηση της απάτης που διαπράτεται κατά των πολιτών. Θα ήθελα τέλος να αναφέρω δύο τομείς στους οποίους αναλαμβάνουμε δράση έχοντας κατά νου την ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων. Στο λιανεμπόριο θέλω να αναφερθώ λοιπόν που απασχολεί 33 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Στις 31 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε ένα σχέδιο δράσης που επικεντρώνεται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική του αποδοτικότητα. Δουλεύουμε μαζί με τους εργαζομένους στον τομέα αυτό για να μπορέσουμε να άρουμε τα βασικά εμπόδια στην ανάπτυξη αυτού του τομέα και ακριβώς αυτές είναι, αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις και να δημιουργήσουν ε, ε, φραγμούς στα σύνορα που θα είναι εις βάρος της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς αυτού του κλάδου ξεκινώντας από τη δράση μας αυτή από τις αρχές του έτους. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, και πάλι θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών με την οδηγία που έχουμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, με την επίλυση διαφορών, ε, με τις δυνατότητες σύγκρισης τιμών και θα προτείνουμε και μια αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις πληρωμές ούτως ώστε να μπορούμε να δράσουμε υπέρ των εμπόρων και υπέρ των καταναλωτών. Θα καλύψουμε και θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού και προστασία δεδομένων. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι και για μένα και για όλους ε, τους ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους άλλους επιτρόπους, γιατί δεν είμαι εγώ μόνος ενδιαφερόμενος. Αυτή η οδηγία παραμένει προτεραιότητα για μας. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική ε, εργασία για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλες οι σχετικές διατάξεις. Έχοντας επισκεφθεί τις πρωτεύουσες των κρατών μελών και έχοντας συναντήσει υπαλλήλου στα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνοι για τα νομικά αυτά κείμενα, χρειάζεται, βλέπουμε, ένας επικοδομητικός διάλογος με τα κράτη-μέλη να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται είτε αρνητικά είτε θετικά σε αυτό το χώρο. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα στο πλαίσιο του διαλόγου που έχουμε με το, την Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου και με τον πρόεδρο Μάρκον Χάρμπορ να σας καλέσω να συμμετάσχετε στο μήνα ε, για την εσωτερική αγορά που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας διάλογος που γίνεται ε, online και περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Ε, έχουμε ανοίξει μια πλατφόρμα σε 24 γλώσσες για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες και θα ασχοληθούμε με το εμπόριο online, με τις τράπεζες, με διάφορα θέματα τα οποία αφορούν άμεσα και την οδηγία για τις υπηρεσίες. Τέσσερις εβδομάδες λοιπόν διαλόγου που θα μας βοηθήσουν να, δούμε πώς αυτή η οδηγία μπορεί να εξυπηρετήσει την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Επιτροπής Απασχόλησης, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κατά αυτή την περίοδο τη τόσο μεγάλη ε, ανεργίας στα κράτη-μέλη, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό το πώς εμεί θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλε τι δυνατότητε τη ενιαίας αγοράς βοηθήσουμε να υπάρξει ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία. Ακριβώ λόγω τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα και συγκύρωση στα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι σχετικέ ε, αλλαγέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο στην εισηγήτρια για το έργο το οποίο επιτέλεσε. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι έχουμε κάποιες πτυχές της ε, γνωμοδότησης από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που αγκάλιασε αυτή η έκθεση. Επίσης, ε, έχουμε αυτά τα σημεία της ενιαίας θηρίδας, ενιαίας επαφής, οπότε είναι πάρα πολύ αυτό το ότι αναφέρεται η ενιαία ψηφιακή αγορά και επίσης το ότι θα πρέπει να τηρηθεί, να εφαρμοστεί η οδηγία. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε την ενεργεία, να ολοκληρώσουμε αυτή την ψηφιακή ενιαία αγορά. Τέλος δε, με μεγάλη μου ε, χαρά βλέπω ότι πρόκειται μια σωσμένη έκθεση και εγώ θα την επιψηφίσω ομάδων και πρώτα θέλω να καλέσω στο βήμα την συνάδελφο Γκάλ Πέλτς για δύο λεπτά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Αναμαρία Κοράτσα Μπίλτ, για την έκθεσή της, διότι ε, τα σημεία τα οποία αναφέρει είναι σημαντικά και θα αποτελέσουν την αφετηρία για το μέλλον. Νομίζω ότι η έκθεση ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας, δηλαδή να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια ανοιχτή αγορά για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Είναι διαφορετική εικόνα που παρουσιάζεται και σύμφωνα με αυτό που είπε και ο κύριος Μπαχνιέ, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να έχουμε μία στο δυνατόν περισσότερο ομοιογενή κατάσταση. Η ανάλυση και τα αποτελέσματα των αναλύσεων ε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε συστάσεις οι οποίες θα είναι διαφορετικές αναχώρα και στόχος ε, της οδηγίας είναι να αρθούν τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις. Για μένα ως πολιτικό είναι επίσης σημαντικό οι ε, εκλογείς μας ε, να μπορέσουν να εκτιμήσουν το ότι η αγορά είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να μπορέσουν να ασκήσουν κάποια δραστηριότητα. Θέλουμε η ενιαία αγορά να μην δρά ως φραγμός αλλά ως κινητοποίηση για τις ε, επιχειρήσεις και αυτό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για άλλες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εναρμόνιση. Ξέρω ότι Ήδη έχουμε πει πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για να υποστηρίξουμε την αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τις ε, υποστηρίξουμε. αν μπορέσουμε να βρούμε καινοτόμε λύσεις ε, θα μπορέσουμε ε, να στηρίξουμε και την ισορροπία που πρέπει να επικρατήσει στον τομέα. Καινοτόμε λύσεις που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι πολίτες της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η συνάδελφος Ιβάνα Ράπτη από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την καλή συνάδελφο την κυρία κοράτσα μπιλτ για τη δουλειά της. Ε, ωστόσο ε, έχουμε ορισμένα σημεία που πρέπει εδώ να επισημάνουμε. το πρώτο σημείο είναι ότι εργαστήκαμε καλά και κάναμε πολύ σκληρές προσπάθειες για να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο συνεννόησης. μέχρι ένα σημείο το καταφέραμε. το αποτέλεσμα ήταν από την πλευρά των σοσιαλιστών να δώσουμε τη συμβολή μας σε τέσσερα σημεία ειδικότερα έγινε σαφές ότι η αναφορά σε ανάπτυξη μέχρι δύο έξι σε μια περίοδο πέντε δέκα χρόνων είναι μια πολύ φιλόδοξη διατύπωση με αρκετές δυσκολίες πραγματοποίησης γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. δεύτερον ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για διασταλτική και πέρα από το γράμμα της οδηγίας ερμηνεία τονίσαμε ότι όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές συνθήκες σε κράτος μέλος. και τέταρτον ισορροπήσαμε την υπερβολική κριτική της έκθεσης στις εθνικές ρυθμίσεις. υπάρχει όμως ένα σημείο ένα σημείο κομβικό για μας τους σοσιαλιστές που είναι το θέμα της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων έτσι ακριβώς όπως το ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος μπαρνιέ. γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες στην ολομέλεια ειδικότερα δε η τροπολογία με τον αριθμό 2 και η τροπολογία με τον αριθμό πέντε που αναφέρονται στην οριζόντια κοινωνική ρήτρα και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων για μας είναι κόκκινη γραμμή. ακούγοντας και τον κύριο μπαρνιέ καλό και τώρα εδώ στην ολομέλεια την καλή συνάδελφο κυρία κοράτσα μπιλτ να υποστηρίξει αυτές τις τροπολογίες οι οποίες στηρίζονται ακριβώς στη γνωμοδότηση του καλού της συναδέλφου του κυρίου Κάζα από την επιτροπή απασχόλησης. θα είναι για το καλό όχι του κοινοβουλίου όχι της ευρώπης αλλά των πολιτών και των εργαζομένων στην ευρώπη. έτσι θα δώσουμε πραγματικά ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτό που λέμε ενιαία αγορά και που την έχουμε ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ράπτη. Ο συνάδελφος Μάλκομ Χάρμπορ από το ECR. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με χαροποιεί ιδιαίτερα η έκθεση αυτή και όπως ανέφερε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ είναι η τελευταία μία σειρά εκθέσεων που παρουσιάζει ε, αυτή η Επιτροπή στην Ολομέλη και στο ευρύτερο κοινό για να τονίσει πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνηση έτσι ώστε να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες καθώς και το ρόλο που παίζει στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Απελπισμένα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και είναι σαφές ότι οι αυξανόμενες υπηρεσίες χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους, περισσότερο γρήγορα από ότι οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. Και αυτό είναι κάτι που έχουν σαφώς δείξει οικονομικές αναλύσεις εδώ και χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι επίσης σαφές ότι οι υπηρεσίες έχουν, ε, ενεργοποιούν την οικονομία. Υπάρχουν πολλοί τομείς που χρειάζεται περισσότερη πραγματο... Ε, περισσότερες ικανότητες στον τομέα του σχεδιασμού κτηρίων, στον τομέα του προγραμματισμού. Όλες αυτές είναι υπηρεσίες και τομείς όπου χρειάζεται περισσότερος ενεργός ανταγωνισμός. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν ήμουν επικεφαλής της ε, αποστολής στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Το ότι ακούσαμε από τα συνδικάτα για την έλλειψη ανταγωνισμού ή ανταγωνιστικότητα στην, ευρωπαϊκή, στην ελληνική οικονομία. Και ακούσαμε από το Υπουργό Ανταγωνιστικότητας να μας λέει πώς το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα επικεντρώθηκε στο ρόλο των υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι που ισχύει παντού συνάδελφοι και θα πρέπει να επιληφθούμε. Πολύ σωστά η κυρία Ράπτη ότι χρειαζόμαστε θεμητό ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν οι θέσεις και οι οικονομικές δραστηριότητες που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Obrigado, Presidente. Esta é uma história com alguns anos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 να οδηγήσουν σε μια, σε, και να πλήξουν τα, ε, τους μισθούς και τα ημερομίστια. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες, δυσκολίες που τους υποχρεώνουν να επιβραδύνουν για παράδειγμα, η οδηγία για τι υπηρεσίε το 2006 οδήγησε σε πολλέ διαδηλώσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι που οδήγησε και σε ευρωπαϊκές διαδηλώσει. Διαδηλώσει που απέρριπταν το άνοιγμα την αγορά σε χώρες όπου το κράτος έπαιζε κοινωνικό ρόλο μέσω δημοσίων υπηρεσιών. Διαμαρτυρίε συγκεντρώσει που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε στο μέλο και που η είναι κατά ε, της ε, διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός είναι ένας τομέας που πλήττεται για να μπορέσουν να αναλάβουν έργα μεγάλες οικονομικές ομάδες, μεγάλη οικονομική ε, όμιλη. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. <laughs> Περνάμε στους ε, υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές και ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μάζε Κούκοβιτς. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και την εισηγήτρια αλλά και τον κύριο Επίτροπο. Μιλούμε τώρα για κάποια συγκυρία που έχει φέρει πάρα πολύ ψηλή ανεργία και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να περιχαρακώσει κανείς τις υπηρεσίες, μια νέα αγορά γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξουν κάποιες λύσεις, πώς οι λύσεις αυτές θα υλοποιηθούν. Ε, είναι κάποιες λύσεις που έχουν δοκιμαστεί αλλά δεν τηρήθησαν στο παρελθόν. Θα πρέπει επομένως να δούμε πώς σε πάρα πολλέ χώρες του ευρώ ε, κάποια βήματα που γίνονται δίνουν κάποια ακτίδα ελπίδας θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε λιγότερο μεταξύ μας και περισσότερο με άλλες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινθία, η Κίνα. Επίσης ε, έχουμε και άλλη μία μια ε, ε, πρόκληση όπως η ΜΜΕ και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ευκολότερη προσβασιμότητα στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι εύκολο γιατί το κάνουμε μεγάλες εταιρείε, αλλά οι μικρότερες είναι πιο δύσκολο. Η ψηφιοποίηση επίσης μας δίνει μια άλλη διάσταση της από απόστασης δράσης στην ενιαία αγορά. Έχουμε βέβαια τα προϊόντα απομίμησης που μας δημιουργούν ε, πάρα μεγάλη απεσιοδοξία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε την νομοθεσία, πώς θα έχουμε κάποια συνέπεια στις, στα πρώτα που αγκαλιάζουμε, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κυρίως να ωφεληθούν από αυτό η νέη η γενιά του ιντερνετ, επίσης η γύρανση του πληθυσμού, ε, προσφέρει κάποιες ευκαιρίες γιατί έχουμε τώρα τις κατοίκων από απόσταση υπηρεσίες. Όσο όλα αυτά τα προωθούμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα 27 εκατομμύρια των ανέργων Ευρωπαίων ε, θέλουμε ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τα 5 εκατομμύρια των νέων ανέργων. Οπότε σίγουρα η εσωτερική αγορά είναι ένα εργαλείο παρακολουθήσιμο για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Μπαχνιέ, αναφέρετε ήδη ότι ήδη έχουν συνταχθεί πολλές εκθέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Από τις προηγούμενες αυτές τις εκθέσεις, σε καμία δεν είχαμε τόσο συμπυκνωμένη την κοινωνική ε, διάσταση της αγοράς με τόσο αρνητικό τρόπο όπως αυτή την οδηγία. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ο έπαινος του εκπροσώπου της Επιτροπής Απασχόλησης διότι από τις τροπολογίες που συντάχθηκαν καμία δεν έγινε αποδεκτή στην ΙΜΚΟ. Νομίζω ότι κάποια διόρθωση πρέπει να γίνει. Στο άρθρο 1 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες υπάρχει υποχρέωση για την κοινωνική διάσταση. Και στην συνθήκη της Λισαβόνας ε, αναφέρεται ότι μιλάμε για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και όχι για μια φιλελεύθερη οικονομία της αγοράς. Και αυτό πρέπει να εκφράζεται σε ένα τέτοιο κείμενο. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, αν αύριο δεν γίνει κάποια διόρθωση υπό αυτή την έννοια στις ψηφοφορίες, η πολιτική μας ομάδα δεν θα είναι σε θέση να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης αυτής. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε κατά παρότι για μας η εσωτερική αγορά είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και παρότι για μας αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει για τις υπηρεσίες είναι κάτι που θέλουμε να εφαρμοστεί. Αλλά δεν μπορούν να δεχθούν οι σοσιαλιστές και δημοκράτες μια τέτοια οδηγία. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Καστέξ δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι ε, η απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο ε, είναι ένας από τους πολλαπλούς, ένα από τα πολλαπλά χαρακτηριστικά του, του τομέα. Αυτό υπήρχε ήδη από την οδηγία Bolkenstein. Υπάρχουν πολλές φορές ιδεολογικές φορτίσεις και πολύ συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως ο κοινωνικός τομέας. Και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου έγινε προσπάθεια να διορθώσουμε κάποια κενά. Δεν μπορεί να απελευθερωθεί η εσωτερική αγορά μόνο με διατάξεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, και οι απαιτήσει των πολιτών. Μία ε, αναζωογόνηση ε, της προσπάθειας που είχε καταβληθεί στο παρελθόν από την πίσω πόρτα δημιουργεί προβλήματα χρειάζεται μια ε, σταδιακή, ένα σταδιακό άνοιγμα του κοινωνικού τομέα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφέ, πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική έκθεση όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη σχετική οδηγία. Έχει να κάνει επίση με το πώ θα δώσουμε νέο δυναμισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία, πώ θα άρουμε κάποιου φραγμού, κάποιο είδου ε, εμπόδια γραφειοκρατικά. Οπότε άκουσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει το θέμα τη ε, δυσμενή διάκριση βάρο των καταναλωτών επί τη βάση τόπου διαμονή και εθνικότητα. Γιατί και στην πράξη όντω έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πρόκειται ε, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην εσωτερική αγορά. Πάντως έχουμε τη γεωνική διάσταση της αγοράς αυτής που είναι πολύ σημαντική και επίσης ε, έχει να κάνει με το βιβλικό επίπεδο, τις συνθήκες απασχόλησης και όταν μιλούμε για γεωνική πρόνοια, ε, για προστασία στην αγορά. Δηλαδή τελικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Ραπτή και τους άλλους προλαλήσαντες. Συμφωνώ κύριε Επίτροπη μας και θέλω πρώτα να παρακαλέσω την συνάδελφο Μάλετιτς να πάρει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την άριστη εκθεσή της. Το να αναβαθμίσουμε την εσωτερική αγορά υπηρεσιών είναι το κλειδί για την πολιτική μας ενόψη του 2020. Θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και την απασχόληση. Έχουμε τον ε, προπολογισμό μας, ο οποίος είναι το εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε καλύτερα ε, την, την πολιτική μας για την αγορά υπηρεσιών. Επίσης, έτσι μπορούμε να άρουμε τα διοικητικά και τα άλλα ε, εμπόδια και τους φραγμούς που έχουμε, ώστε να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες και έτσι μπορέσουμε να έχουμε πιο εύρυθμες διοικητικές διαδικασίες για την παροχή των υπηρεσιών και έτσι επίσης θα έχουμε μια αυθεντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ο τομέας των υπηρεσιών ε, είναι το 70% του ΕΕΠ των κρατών μελών. Είναι το κλειδί, είναι κομβική σημασίας για το πώς θα βοηθήσουμε την απασχόληση, για το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό εισόδημα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε την ε, πιο αρμονική αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων. Αυτό έχει να κάνει ε, φυσικά με την αγορά των υπηρεσιών. Επίσης συζητήσαμε και το τόσο δυνερό θέμα της ανεργίας των νέων πάνω από 90%. Μία από τις λύσεις, όπως το λέει και η έκθεση, είναι το να ανοίξουμε κάποιες θέσεις απασχόλησης της υπηρεσίας. Να συμμετοχθούν αυτή την ευκαιρία. Θα καλέσω να κάνετε μία προσπάθεια να τηρείτε το χρόνο σας. Τσέντζο, Κοφεράτη. Grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα το παρουσιάσατε εσείς. Μας θυμίσατε ότι στην εφαρμογή της οδηγίας επί των υπηρεσιών σε πολλές χώρες παρατηρούνται καθυστερήσεις ή παραλήψεις. Δεν πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο πεπρωμένο τους. Το γεγονός είναι ότι την οδηγία αυτή τη σκεφτήκαμε σε μία φάση ανάπτυξης και η κρίση που επήλθε αργότερα άλλαξε τις αντικειμενικές συνθήκες της εφαρμογής της. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να καταλήψουμε το στόχο μας. Όχι, θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Θα πρέπει όμως να αλλάξουμε τους χρόνους. Ε, δεν μπορούμε ε, να κάνουμε αυτό που φανταστήκαμε αρχικά. Το δεύτερο θέμα αφορά την κοινωνική διάσταση των δράσεών μα. Ε, η οριζόντια ρήτρα, η οριζόντια κοινωνική ρήτρα είναι αναγκαία όχι μόνο για τα άτομα που εργάζονται αλλά και για τι επιχειρήσει. Εάν δεν υπάρχει ένα ενιαίο κατόφλι παγκόσμιο, ο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που επικοδικοποιούνται γίνονται διαγράφοντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώ αυτή είναι η χειρότερο ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει στον κόσμο και αυτό είναι σημαντικό αυτή η διάθεση και κυρίω το να αποκτήσει ένα χαρακτήρα, έναν ε, ναι, ενιαίο χαρακτήρα αυτή η κοινωνική διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κοράτσα για τη θαυμάτισια δουλειά που έκανε. Είμαι σίγουρη ότι αυτό αποτελεί ένα μοχλό για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης. Η εφαρμογή αυτής της αγοράς θα μπορούσε να φτάσει στο 2,6% του ΕΠΑ. Αυτό επιβάλλει ότι θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, ένα σοβαρότερο εμπόδιο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά να μειωθούν και οι πρακτικέ διάκριση που έχουν άμεση επίπτωση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Συμφωνώ με την ανάγκη του να υπάρχει αλληλεπίδραση με την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα, γιατί θα ήταν σκόπιμο οι χώρε μέλη να καταργήσουν τις ε, ανώφελες, ε, ε, τα ανώφελα πετούμενα για την πρόσβαση σε ένα επάγγελμα. Στη χώρα μου υπάρχουν πολλέ οδηγίε στη χώρα μου, η χώρα μου πάσχει για παράδειγμα για διακρίσεις που γίνονται σε ορισμένους τομείς. Θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και για το λόγο αυτό θα καλούσα για μία ακόμα φορά να επισκεφτεί τη χώρα μας και να μας βοηθήσει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή λείπει εντελώ η προβληματική που αφορά την εφαρμογή τη οδηγία υπηρεσιών σε διάφορε χώρε μέλη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομεί, κατηγορίε εργαζομένων που διατρέχουν το κίνδυνο να βρεθούν χωρί απασχόληση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στου Ιταλού ε, που εργάζονται, ε, ε, που είναι ανταπαραίτητο επάγγελμα. Αναρωτιέμαι γιατί θέλουμε να θυσιάσουμε επηρεάσουμε αυτή την κληρονομιά για να αφήσουμε περιθώριο σε μεγάλες ε, τουριστικές επιχειρήσεις που απλά και μόνο θέλουν να αφήσουν το σημάδι τους ε, στι ακτέ μα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι υπέρ τη ευρωπαϊκής οικονομίας και των πολιτών. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι ε, ωφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν σε μια απελευθέρωση των τυπικών προσόντων για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, οι ξεναγοί, που καλούνται να επιδείξουν την ιστορική μας κληρονομιά που είναι μοναδική στον κόσμο. Προέρχονται από μια πάρα πολύ αυστηρή εκπαίδευση η οποία στόχο έχει να δώσει, δείξει το καλύτερο της πρόσωπο σε όλους τους τουρίστες. Υπάρχουν χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες που πιστεύω ότι θα πρέπει να τύχουν κάθε σεβασμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, κυρίους και κυρίες βουλευτές που εκφράστηκαν ε, σαφέστατα για να προσπαθήσουν να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις που όμως όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν την Επιτροπή στο να διαρωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος μας ε, και τι πρέπει να κάνουμε για να εφαρμόσουμε αυτήν την οδηγία. Και αυτή την οδηγία και όλες τις άλλες οδηγίες που εσείς έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν για τις υπηρεσίες με έναν τρόπο έξυπνο και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με το θέμα ε, των ακτών. Ε, είναι κάτι το οποίο ε, έχει περάσει μέσα στο κείμενο της οδηγίας και εμείς πρέπει να το εφαρμόσουμε και γι' αυτό το κάνουμε με τον πιο έξυπνο τρόπο, με τον πιο επικοδομητικό τρόπο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε επιτόπου αυτές τις διατάξεις ενώ ταυτόχρονα θέλουμε και να ενισχύσουμε την τουριστική δραστηριότητα στις ακτές της Ιταλίας. Ε, τώρα προς τον κύριο Φερέιρα καταλαβαίνω τις ανησυχίες ε, σε σχέση με αυτήν την οδηγία και τις υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο αποδυνάμωσης ε, υπηρεσιών που προηγουμένως παρήχε το κράτος. Η οδηγία στην οποία συνεισφέρεται τόσο πολύ πριν από λίγα χρόνια ήταν μια οδηγία διοικητικής απλούστευσης και οι κοινωνικές υπηρεσίες εν μέρη καλύπτονται. Εξάλλου το Κοινοβούλιο είχε απορρίψει μια τροπολογία για τον αποκλεισμό αυτών των υπηρεσιών. Αν παρέχονται όμως από το κράτος αυτές οι υπηρεσίες αποκλείονται από το πεδίο Όσον αφορά τις υπηρεσίε ε, γενικού ενδιαφέροντος, ε, ε, είναι ένα τομέα στο οποίο δεν εφαρμόζεται η προσωρινή παροχή αυτών των υπηρεσιών διαμεθοριακά. Πολλοί αναφέρατε την ε, κοινωνική προστασία, την προστασία των εργαζομένων και θέλω να πω ότι η οδηγία, όπω εγώ τη διαβάζω, όπω εγώ την καταλαβαίνω και όπω εγώ θέλω να εφαρμοστεί, είναι σαφέστατη για αυτό το θέμα. Δεν επηρεάζει το εργατικό δίκαιο, δεν επηρεάζει το δικαίωμα διαπραγμάτευση, το δικαίωμα σύναψη συλλογικών συμβάσεων, ούτε το δικαίωμα συλλογικών δράσεων. Ειλικρινέστατα ε, δεν γνωρίζω να έχει παραβεί κάποιο κράτος μέλος την οδηγία όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να παίξουν παράλληλα με εσάς ένα σημαντικό ρόλο να φροντίσουν ώστε να λαμβάνονται μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να υλοποιείται η οδηγία αυτή για τις υπηρεσίες τηρώντας ε, σε όλα αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα από την ε, έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ ε, που είναι εμπεριστατωμένη και δυναμική εγώ παίρνω ένα βασικό μήνυμα που απευθύνεται και σε μένα και στα κρατημέλη να φτάσουμε πραγματικά μέχρι τέλους αυτή την οδηγία να της δώσουμε ε, όλες τις δυνατότητές της, γιατί ξέρουμε ότι έχει δυναμικό ανάπτυξης ε, της οικονομίας στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να αρκεστεί στο να είναι μια οικονομία υπηρεσιών. Θα πρέπει να αναζητήσει τη φιλοδοξία ε, του να είναι μια βιομηχανική δύναμη, μια παραγωγική δύναμη. Αλλά τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα, στον τομέα των υπηρεσιών που συζητάμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση αυτή τη οδηγία με, όλο, ε, με όλες δυνατότητες που μας δίνει. Και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε αυτή την οδηγία με μηδενική ανοχή και εμείς και τα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία επ' αυτού. Αυτό εντάσσεται στην οικονομική γραμμή την οποία ακολουθούμε. Ποτέ δεν έχουμε εγκαταλείψει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μερικές φορές μπορεί μια γραμμή να την έχουμε εγκαταλείψει λίγο στις οικονομικές αγορές, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς και αυτές ε, οι λέξεις είναι όλες σημαντικές, ε, όχι λίγες από αυτές τις λέξεις, αλλά το πλήρες νόημα της φράσης. Ευχαριστώ. Κομισέρ. Ευχαριστούμε. Συγγήτριά μας, την ε, συνάδελφο Κοράτσα Μπίλτ για τα καταληκτικά της σχόλια. Thank you very much, uh, Madam Chair. We appreciate all colleagues' comments. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Καταλαβαίνω ότι διαφορά στις ευαισθησίες που υπάρχουν και την ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση στις χώρες μέλη. Βεβαίως ο καλύτερος τρόπος για να συμπεριληφθεί η κοινωνική διάσταση είναι το να διασφαλίσουμε μια θέση εργασίας για όλους. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι με τη δουλειά τους μπορούν να φροντίσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Η οδηγία αυτή συμπεριλαμβάνει, όπως είπε η κυρία Γκάρο, στο άρθρο 1, την κοινωνική διάσταση και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η συνδική τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται να επαναληφθεί για μία ακόμα φορά. Θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Όλοι είμαστε υπέρ αυτή. Εδώ έχετε δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι πραγματιστική αυτή που πρόβαλε ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Ας κοιτάξουμε τους περιορισμούς, ας κοιτάξουμε τα προβλήματα, ας δούμε πόσο απτά μπορούμε να συνεργαστούμε με τις χώρες μέλη έτσι ώστε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την, ε, τα εμπόδια. Υπάρχει μια ιδεολογική θέση που λέει ας επαναλάβουμε χιλιάδες φορές τα όσα συμπεριλαμβάνονται ήδη στα κείμενα για να τονίσουμε ότι εμείς είμαστε υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ε, ε, την κυρία τη συνεργαστήκαμε στενά και πραγματικά με πλήσει την Ολομέλεια αφού έχουμε πραγματικά καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνουν όλοι οι συμβιβασμοί που να είναι ικανοποιητικοί για τις ομάδες κόκκινε, τι πράσινες. Έρχεστε εδώ τραβώντας συγκεκριμένες γραμμές και απειλώντας. Δεν καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να απολογηθείτε στους λαούς της Ευρώπης, όχι σε μένα. Ζητάω την άδελφη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα στις χώρες μέλη έτσι ώστε θα κρατηθεί σε υψηλότερο επίπεδο στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μπορέσουμε να άρουμε τα εμπόδια για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά υπηρεσιών, για να υπάρχουν θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα. Μην την αμβλύνετε, ας στρέψουμε το βλέμμα στο αύριο και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, απόλυτα την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κοράτσα Βίλντα. Συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία για την ε, έκθεση της συναδέλφου Κοράτσα Μπίλ θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη.